Chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Καλημέρα. Θα ήθελα να σας ζητήσω να καθίσετε και σας καλωσορίζω τόσο νωρίς σήμερα το πρωί για την τελική συνεδρίαση της, ε, των δύο επιτροπών μας, Οικονομικών Υποθέσεων και Προϋπολογισμού. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, στρατηγικών επενδύσεων για την παράταση αυτό. Δεν έχουμε παρατηρήσει για την σε διάταξη, οπότε εγκρίνεται. Θέλω να ε, παληθέσω αν εγκρίνεται τα πρακτικά της κοινή συνεδρίασης που έγινε στις 15 Μαΐου 2017. Αυτά τα πρακτικά λοιπόν εγκρίνονται. 26 Οκτωβρίου η διοργανωτευτική ομάδα Badge Econ έφτασαν σε πολιτική συμφωνία με την Εστονική Προεδρία του Συμβουλίου όσον αφορά την παράτωση της διάρκειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων του ΕΤΣΕ. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε ε, μία ε, επιστολή της 8ης Δεκεμβρίου ότι το Κορεπέρ δεχόταν αυτή την πολιτική συμφωνία. κάναμε τις διαπραγματεύσεις λοιπόν με το Συμβούλιο και υιοθετήθηκε η πρόταση στις 15 ε, Μαΐου. Η επιστολή της Κορεπέρ καθώς και το κείμενο της συμφωνίας έχουν διαβιβαστεί στα μέλη των Επιτροπών μας στις 9 Νοεμβρίου ε, εν ώψη της νέας διαβούλευσης σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με το άρθρο 69F4 του κανονισμού Badge Econ, τώρα θα ψηφίσουμε επί τη βάση της προσωρινής πολιτικής συμφωνίας, αλλά υπάρχει μια διευκρίνηση διαδικαστικού τύπου και ε, δίνω το λόγο στο σύμπροεδρο Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη. Ευχαριστώ, Ζαν. Θέλω να κάνω την εξής ε, δήλωση. Υπάρχει ένα ε, τυπικό λάθος στην παράγραφο 9.2.1α νέο στην παγιωμένη εκδοχή της συμφωνίας που συνοδεύει την επιστολή Κορεπέρ ε, και επιβεβαιώθηκε χτες, ε, λάβαμε επιβεβαίωση από την Προεδρία ότι θα επικυρωθεί αυτό το κείμενο ε, πριν από την ψηφοφορία στην Ολομέλη. Είναι η στάνταρ πρακτική και το κείμενο λοιπόν λέει ενώ αναγνωρίζουμε το αίτημα για την παράταση του ΕΦΣΙ, η οποία θα στοχεύσει τουλάχιστον στο 40% της χρηματοδότησης του ΕΤΣΕ, υπο, τις υποδομές ε, και την ε, καινοτομία που στηρίζει τμήματα project που θα συμβάλλουν κτλ. Πρόκειται για μια τεχνική σε φύσης διόρθωση και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι εξαιρετικά περήφανοι και ικανοποιημένοι για το, ε, την έκβαση των διαπραγματεύσεων. Είχαμε εξαίρετη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών μας, μεταξύ των εισηγητών, μεταξύ των σκιωδών και του μεγάλου αριθμού πολιτικών ομάδων που συνέβαλαν στη σημαντική βελτίωση του κειμένου και θα δώσω το λόγο στους δύο εισηγητές για σύντομες ε, παρεμβάσεις. Παρακαλώ. Ναι, πολύ σύντομος. Σας ευχαριστώ. Και ευχαριστώ το Προεδρείο της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμού και της Επιτροπής ε, Οικονομικών ε, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή Μπούλμαν. Κάναμε εξαιρετή δουλειά, πιστεύω, και τους στόχους που είχαμε εξαρχίσει τους καταφέραμε στο τέλος. Βεβαίως και ευχαριστώ και όλους τους σκιώδεις εισηγητές. Όταν το κυροβούλιο είναι ενωμένο, καταφέρνει να επιτύχει τους στόχους του. Πολύ σύντομα. Γλιτώσαμε 225 για το ΣΕΦ, Connecting Europe Facility. Ε, το Συμβούλιο ε, δεν ήθελε το Συμβούλιο τα 150 εκατομμύρια για την εισεγγυήσει από την ε, αναδίπλωση. Λάβαμε φρέσκο χρήμα και μετά έχουμε τώρα έναν κανονισμό όπου ενισχύσαμε την προσθετικότητα, την παρουσία του Κοινοβουλίου και την διαφάνεια. Παρουσία του Κοινοβουλίου, για παράδειγμα, στο Steering Board, στο Διοικητικό Συμβούλιο, με ορισμό κάποιου ε, συν ε, περισσότερη λογοδοσία δηλαδή. Οι λιγότερο ανεπτυγμένες ε, περιφέρειες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν περισσότερο γιατί εκεί έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή των National Promotional ε, ε, και μετά έχουμε την συμβουλευτική πλατφόρμα ε, και μετά θα έχουμε έτσι μια πιο δραστήρια στάση. Είμαστε στο καλό δρόμο. Ελπίζω πως η ΕΤΕΠ θα ερμηνεύσει καλά τον κανονισμό για περισσότερη ανάπτυξη, περισσότερη απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως απασχόληση για τους νέους σε όλες τις περιφέρειες, με μια σωστή, ωραία ε, γεωγραφική ισορροπία και επενδύσεις που θα πρέπει να είναι βιώσιμες, αλλά και φιλικές προς το περιβάλλον, διότι ενισχύσαμε και το ζήτημα του κλίματος και τους στόχους του κλίματος. Ευχαριστώ όλους και είμαι βέβαιος ότι θα πάει καλά το πράγμα. Κύριος Μπούλμαν, ευχαριστώ τους δύο συμπροέδρους. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Χωσέ Μανουέλ. Ήταν πραγματικά ομαδικό το έργο μας. Θέλω όμως να ευχαριστήσω και όλους τους ε, σκιώδεις εισηγητές από τις ε, δύο επιτροπές και θα ήθελα ιδίω σήμερα να συγχαρώ και τα επιτελεία της ομάδας των ανθρώπων που εργάζονται πίσω από τους ευρωβουλευτές και τους υποστηρίζουν και που επίσης επιτέλεσαν εξαιρετικό έργο. Τι είναι το, ποιο είναι το σημαντικότερο επίτευγμα του Κοινοβουλίου όσον αφορά το έτσι 2. Είστε όλοι σας έμπειροι πολιτικοί, αγαπητοί συνάδελφοι. Και γνωρίζετε αυτήν την διοικητική λογική. Πότε μπορεί να χαρακτηριστεί ένα πρόγραμμα ως αποτελεσματικό. Η απάντηση είναι όταν έχουν αξιοποιηθεί όλα τα κονδύλια που διέθετε το εν, το λόγω πρόγραμμα. Ε, αυτήν τη λογική την έχουμε διαρρήξει πλέον. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει πλέον δεν είναι απλά να απορροφηθούν τα κονδύλια, να δαπανηθούν τα χρήματα, αλλά να μπορέσουμε να επιλύσουμε προβλήματα στις περιφέρειες, να εξυγχρονίσουμε την, την οικονομία μας, να γίνουν απαραίτητες προσαρμογές, αλλά αλλαγές που θα έχουν νόημα. Να μην κρίνεται η επιτυχία ενός προγράμματος μόνο από το κατά πόσο δαπανήθηκαν τα κονδύλια, αλλά από την ευρύτερη λογική και την πλαισίωση του προγράμματος. Και αυτό το έχουμε επιτύχει. Περισσότερη ποιότητα, περισσότερη διαφάνεια, συμπληρωματικότητα, διακυβέρνηση με διαφανή τρόπο που καταδεικνύει πού κινούνται και προς τα πού πηγαίνουν τα πράγματα και έτσι το έτσι θα καταστεί ένα υψηλής ποιότητας προϊόν που έχει δημιουργηθεί εδώ στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτή είναι η επιτυχία μας. Η επιτυχία μας αυτή, όπως είπε και ο Χωσέ Μανουέλ, κατέστη δυνατή ακριβώς γιατί συνεργαστήκαμε πέρα από κομματικά στενά όρια. Και όλα αυτά χωρίς να παρεκκλίνουμε καθόλου από την αρχική εντολή του Κοινοβουλίου. Έγιναν διαπραγματεύσεις για όλα τα θέματα σε βάθος. Και αυτό είναι κάτι που λείπει και από το Κοινοβούλιο, πρέπει να σας πω με ειλικρίνεια. Ήταν ε, λοιπόν μια εξαιρετική διαδικασία που νομίζω ότι μπορεί να δράσει και ως ε, υπόδειγμα για το πώς μπορούμε να, να αξιοποιήσουμε... Ε, τέτοιου είδους ευκαιρίες και στο μέλλον. Και νομίζω ότι και στο μέλλον ακριβώς στην Ευρώπη θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να προχωρήσουμε με τον τρόπο που προχωρήσαμε εδώ. Λοιπόν, ωραία, λέει ο πρόεδρο να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία για να περάσουμε στην κανονική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ για να δούμε αν λειτουργούν τα μηχανήματα. Still some colleagues to vote for the test. Problems? Yes, we give you the time. No, now is a test. Τώρα κάνουμε δο δοκιμαστική ψηφοφορία για να δούμε αν λειτουργούν τα μηχανήματα. Some machine not working. Υπάρχουν κάποια μηχανήματα που δεν λειτουργούν. Μπορείς, Φίλιπ, να δοκιμάσεις το άλλο, το διπλανό. Λειτουργεί αυτό. Ωραία. Τέλεια. Τέλος, λοιπόν, στη δημοστική δοκιμαστική ψηφοφορία. Και πάμε στην κανονική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση επί, ψηφοφορία επί της ε, προσωρινής συμφωνίας. Άρχεται η ψηφοφορία. to vote, but it's not mandatory. So... Δεν ψήφισαν όλοι, αλλά δεν είναι και υποχρεωτικό. Κύριε Κλίνς, υπερψηφίζει ο κύριος Κλίνς. 52 υπέρ, 4 κατά, μία αποχή, μεγάλη πλειοψηφία, ευρύτατη πλειοψηφία, συγχαρητήρια στους συνεισηγητές, εγκρίνεται η έκθεση. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους, στη γραμματεία, στο προσωπικό, στους συνεισηγητές, στους σκιώδεις. Ευχαριστώ, γεια σας.